Good afternoon, colleagues. Καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Βλέπω ναι, ότι κάποιοι δεν είναι εδώ, αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να ξεκινήσουμε. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης πρώτα απ' όλα. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, προτείνω να εγκριθεί με την αλλαγή βέβαια στην ώρα έναρξης, έτσι. Εγκρίνεται η μερίσια διάταξη, συνεπώς. Ε, μια τεχνική ανακοίνωση. Σας ε, υπενθυμίζω ότι η κύρια είσοδος που είναι εδώ δίπλα θα παραμείνει κλειστή για λόγους ευγένεια προς τους προσκεκλημένους μας. Αν τυχόν ε, θέλετε να φύγετε πριν ολοκληρωθεί η συνάντηση με τους προσκεκλημένους μας, παρακαλώ να αποχωρήσετε από τις πόρτες που είναι πίσω. Καλά, όχι από τα παράθυρα, από τις δύο πόρτες που είναι δεξιά και αριστερά. Καλά, Δευτέρα είναι, ο καθένα. Υπάρχουν δύο έξοδοι λοιπόν, εντάξει. Τώρα, σημείο 3 στην ημερήσια διάταξη. Βάσει το άρθρο 204 του κανονισμού, μετά τη συνάντηση των συντονιστών τον Ιανουάριο, ε, φωτώσαμε τα έγγραφα για την ε, συνάντηση στη, στα πρακτικά της σημερινής ε, συνεδρίασης. Σημείο 4 στην ημερήσια διάταξη τώρα, σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Καναδά, κατάσταση πραγμάτων και ποια είναι η κατάσταση μετά από τις εκλογές του Οκτωβρίου. Αγαπητοί συνάδελφοι, Καλωσορίζουμε την Πρέσβερντα που είναι ε, διευθύντρια στην ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπεύθυνη για την Αμερικανική Ήπειρο. Από τις εκλογές του Οκτωβρίου του 2019, το κόμμα των φιλελεύθερων με τον Πρωθυπουργό Τζουστιν ε, Τριντό κέρδισε 157 ψήφους αλλά έχασε την πλειοψηφία που είχε το 2015, την οποία κέρδισαν οι συντηρητικοί που είναι τώρα το κόμμα της αντιπολίτευσης. Έχουμε κοινέ αξίες με τον Καναδά, όπως φαίνεται από τη μακρά ιστορία πολιτικών και οικονομικών ε, σχέσεων και συνεργασίας που έχουμε. Ο Καναδάς είναι μία από τις χώρες εκείνες ε, που είναι περισσότερο ε, φίλοι μας, εταίροι μας από οπουδήποτε αλλού. Είχαμε τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία ΣΕΤΑ, είχαμε τους εισηγητές μας και θα μιλήσουν αν θέλουν. Ο Καναδάς θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά βέβαια μεταξύ μας υπάρχει ωκεανός. Λοιπόν, πέρα από την Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και την Συμφωνία ΣΥΤΑ του 2016, συνεχίζουμε να βαθύνουμε στις σχέσεις μας. Είναι ένας αξιόπιστος εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Καναδάς για θέματα που έχουν να κάνουν με το κλίμα, με τη βιοπικιλότητα, αλλά και παντός είδου συνεργασία στην εξωτερική πολιτική, την πολιτική ασφάλεια, στη τεχνητή νοημοσύνη και την έρευνα. Αυτή η στέρεα εταιρική σχέση θα πρέπει να συνεχιστεί και είμαι πεπισμένος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το νεοεκλεγμένο Καναδικό Κοινοβούλιο θα συνεχίσουν την καρποφόρα συνεργασία και σε αυτή τη θητεία. Αξιότιμοι πρέσβοι, έχετε το λόγο για να μας πείτε πώς βλέπετε εσείς τις επιπτώσεις των πρόσφατων αυτών ομοσπονδιακών εκλογών και τη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά τους επόμενους μήνες. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Εξότιμε πρόεδρε, εξότιμα μέλη της Επιτροπής ΑΦΕΤ, Πολύ χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ μαζί σας και που έχω την ευκαιρία να σας παρουσιάσω περισσότερα για τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε στον Καναδά. Όπως είπατε και εσείς, είχαμε εκλογέ τον Οκτώβριο και η κατάσταση δεν έχει αλλάξει και τόσο πολύ. Άλλαξε, αλλά όπως είπα, όχι τόσο πολύ. Έχουμε λοιπόν τη δεύτερη κυβέρνηση Τριντό τώρα 75% των υπουργών παραμένουν ίδιοι. Δεν περιμένουμε δηλαδή μεγάλες αλλαγές στον προσανατολισμό των πολιτικών μας. Είδαμε το πρόγραμμα της νέας κυβέρνησης και αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το πρόγραμμα αυτό ευθυγραμμίζεται απόλυτα με το νέο πρόγραμμα της Νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό είναι λοιπόν το θετικό Όντω έχουμε μια μακρά ιστορία καλών σχέσεων η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον Καναδά. Όπως επίσης σωστά είπατε, ο Πρωθυπουργό ε, Τριντό είναι επικεφαλής ε, μιας κυβέρνησης μειοψηφία και βασίζεται στην στήριξη άλλων κομμάτων που του υποσχέθηκαν ότι θα τον υποστηρίζουν. Συνεπώς, ε, βγήκαμε αρκετά διχασμένοι από τις εκλογές η κατάσταση είναι αρκετά πολλωμένη ανάμεσα στις επαρχίες ε, του Ανατολικού και του Δυτικού Καναδά, της Υπέθρου και των Πόλων και αυτό το οποίο χρειάζεται τώρα είναι συνοχή και ενότητα. Η κυβέρνηση θα χρειαστεί να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της, ώστε να έχουμε και πάλι ενωμένη τη χώρα. Είναι βέβαια κάτι που βλέπουμε και αλλού στον κόσμο. Ο Πρωθυπουργό θα πρέπει να βρει κοινό τόπο με τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να μπορέσει να προχωρήσει στους ε, στόχους του κατά τη διάρκεια της θητείας αυτής. Πριν από μερικές εβδομάδες, ο Πρωθυπουργό είχε την ομιλία του θρόνου και παρουσίασε τις προτεραιότητες της κυβέρνησή του και το Καναδικό Κοινοβούλιο ενέκρινε τις προτεραιότητες αυτές την Δευτέρα που μας πέρασε, 27 Ιανουαρίου. Οπότε η κατάσταση είναι πιο σαφής και μπορεί να μιλήσει για τις προτεραιότητες. Είναι κλιματική αλλαγή, καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, που είναι το κύριο θέμα για την Ευρώπη και είναι το κύριο θέμα και για τον Καναδά. Ε, μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050. Αυτό είναι που υποσχεθήκαμε. Και επίση υπογραμμίζει η κυβέρνηση και τη φιλοδοξία της να το πετύχει αυτό με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο ώστε να συνεχίζει η ανάπτυξη της οικονομίας και οι τιμές να είναι προσιτές πάντα. Η κυβέρνηση σκοπεύει να υιοθετήσει μέτρα για να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση των κτηρίων και να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μια δεύτερη σημαντική προτεραιότητα είναι οι διαφωνίες που υπάρχουν, διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων επαρχιών να αμβληθούν. Έχουμε και τον Υπουργό Κρίστια Φρίλεν, ο οποίος είναι αναπληρωτής Πρωθυπουργός και υπουργό Διακυβερνητικών Υποθέσεων και θα αποτελέσει την κύρια προσωπικότητα η οποία έχει το σημαντικό ρόλο να διατηρήσει ανοιχτές ε, σχέσεις και συνεργασία μεταξύ όλων των ε, περιφερειών και των ε, επαρχιών. Είναι πολύ κανή και πρέπει να σας πω ότι με ξέπληξε που είδα πόσο πολύ βοήθησε και εδώ στην Ευρώπη με τη Συμφωνία ΣΥΤΑ και πιστεύω ότι θα πετύχει και εδώ. Μία άλλη τρίτη προτεραιότητα της κυβέρνησης τριτό... είναι οι περικοπές που έχει υποσχεθεί, όχι για όλους, για ορισμένους μόνο. Και εδώ το πιο βασικό θέμα είναι να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα για τα φάρμακα Πρέπει να ξέρετε ότι στον Καναδά το σύστημα υγείας δεν καλύπτει τη συνταγογράφηση. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για αυτή την κυβέρνηση. Κάτι άλλο που απορρέει από το προηγούμενο είναι η συμφιλίωση με τους αυτόχθονους πληθυσμούς. Είπε η κυβέρνηση ότι θα τηρήσει πλήρως τη δήλωση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων μέσα στον πρώτο χρόνο μόλις της νέας εντολής. Η φιλοδοξία είναι μεγάλη δηλαδή. Άλλη στόχοι της κυβέρνησης Τριντό τώρα, θα σας τα αναφέρω, είναι η μείωση της ρήπανσης από τα πλαστικά. Αυτό το έχετε κι εσείς εδώ στην Ευρώπη. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό για την Αμερικανική Ήπειρο είναι οι εμπορικές ρυθμίσεις και ε, πρόκειται και για τον αγωγό Trans Εξωτερική πολιτική. Επικύρωση της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών, NCA. Πρόκειται και μια προσυμφωνία ναύτα, που είναι Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Μεξικό. Και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό για τον Καναδά, θα προσπαθήσει να πετύχει μια έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Πρέπει να πω επίσης ότι θα συνεργαστούμε με όλες τις χώρες, ότι ανανεώνουμε τη δέσμευσή μας στο ΝΑΤΟ και την Ειρηνευτική Συμφωνία και θα προσφέρουμε ακόμα μεγαλύτερη βοήθεια βάσει προτεραιοτήτων και επίσης θα εργαστούμε και στο θέμα της εκπαίδευσης και της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων. Κάτι άλλο σημαντικό για την Ευρώπη είναι η αναθεώρηση των κανόνων για τα ψηφιακά, προκειμένου να υπάρχει δικαιοσύνη, να υπάρξουν ε, ε, και ηθικές ε, κατευθυντήριες γραμμές για την ηθική όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα το ακούσατε, όπως σα το είπα και πριν, οι προτεραιότητε μα αυτέ θυμίζουν πολύ τι προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, γνωρίζετε τι είπε η πρόεδρος Φοντερ Λάιεν στο Στρασβούργο τον Νοέμβριο. Μίλησε για τον δρόμο εκείνων που έχει πολλά εμπόδια που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλές αντιθέσεις και ότι θα πρέπει αυτές τις νέες προκλήσεις να τις αντιμετωπίσουμε και ότι αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνο με τους φίλους μας. Ο Καναδάς λοιπόν είναι χώρα που είναι φίλοι μας και ένας πολύ σημαντικός εταίρος για μας. Υπάρχει η συμφωνία SPA, υπάρχει η ΣΥΤΑ που βρίσκεται στο εφαρμοστικό στάδιο και θα θέλαμε φέτος να οργανώσουμε όχι μόνο υπουργική συνάντηση αλλά και διάσκεψη ε, κορυφής με τον Καναδά. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε. προς τα τέλη αυτή της χρονιάς <clears throat> να έχουμε μια τέτοια συνάντηση, τέτοιο επίπεδο. Επίσης, είδαμε μέχρι τώρα και σημαντικές εξελίξεις τα τελευταία χρόνια. Είπαμε για τη συμφωνία ΣΕΤΑ. 10,5% αυξήθηκε ε, το εμπόριο μεταξύ μας σε σχέση με τις προηγούμενες χώρες. Οι εξαγωγές από εδώ αυξήθηκαν 15% και 7% ε, προϊόντα γεωργίας. Όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι είναι σημαντικά. Σε μία εβδομάδα επίσης θα έχουμε την, επιτροπή, την Κοινή Επιτροπή Συνεργασίας που θα αξιολογήσει τις διμερείς μας σχέσεις και θα πρέπει να δούμε αν θα μπορέσουμε ακόμα να οργανώσουμε τέτοιες ε, συναντήσεις, συνεδριάσεις υψηλού επίπεδου ακόμα φέτος. Τι θέλουμε να κάνουμε εκεί, θέλουμε να δούμε επίσης το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε περισσότερα για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τους Καναδούς, για την ισότητα των δύο τη δημοκρατία, το κρατός ε, δικαίου, τη διεθνή τάξη και την ε, πολυμερή προσέγγιση. Επίσης, τι θα κάνουμε με την κλιματική αλλαγή που έτσι καλώς είναι πολύ ψηλά στην ημερήσια διάταξη και ε, στη μία πλευρά και στην άλλη. Θα δούμε επίσης τι δυνατότητες υπάρχουν να προωθήσουμε τις νέες τεχνολογίες. Και βέβαια πώς θα μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη είναι τα ψηφιακά. Είναι προτεραιότητα και για τις δύο πλευρές επίσης, όπως επίσης η ψηφιακή καινοτομία, η τεχνητή νοημοσύνη και θα κοιτάξουμε και την πιο στενή συνεργασία για θέματα ηθικής όταν χρησιμοποιούμε ε, ψηφιακά και γενικά δεδομένα. Ένα άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η ασφάλεια. Υπάρχει συνεργασία ε, για τις ικανότητες που διαθέτουμε για να αντιμετωπίζουμε απειλές και προκειμένου να προωθήσουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα με τη συνεισφορά επίσης του Καναδά σε διάφορες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Ξέρετε ότι ο Καναδάς συμμετέχει στην Ουκρανία για παράδειγμα σε μια τέτοια αποστολή και στο Μαλί και στο Ιράκ. Ο Καναδάς δεν είναι μόνο ένας καλός μας σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, αλλά πριν από μερικές μέρες μάλιστα είχαμε και ένα διάλογο για την ε, ασφάλεια, όπου συζητήσαμε για περισσότερη συνεργασία, τις προτεραιότητές μας και σαφώς είπαμε ότι είμαστε έτοιμοι να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο σε αυτά. Και για να επαναλάβω κάτι που είπατε εσείς, και ακούσαμε και από τον καθηγητή τον Νοέμβριο του 2018 εδώ στην Ευρώπη, καθηγητή ΣΥΡ, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και θυμίζει αυτό που είπατε κι εσείς. Είπε λοιπόν ότι πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένα τα σύνορα της Ευρώπης, αλλά ότι η ότι αν γινόταν κανεί μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει ιδεών και αρχών, τότε ο Καναδά θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μέλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά. Σα ευχαριστώ πολύ. Thank uh, nice... Σας ευχαριστώ πολύ. Τι είναι Καναδός. Ένας άοπλος ε, βορειοαμερικανός χωρίς ασφάλεια. Έτσι, είναι μια άλλη τέτοια που έχω ε, ρίση, που έχω ακούσει για τους Καναδούς. Πιζάπια καταρχάς τώρα, για να έχουμε μία συζήτηση. Ε, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ. Ε, πολύ θετική η παρουσίαση που μας κάνατε. Εγώ έχω, να, έχω δύο ερωτήσεις ε, που προκύπτουν από την πολύ θετική σας παρουσίαση για τις προτεραιότητες οι οποίες είναι παρόμοιες μεταξύ του Ευρωκοινοβουλίου και του Καναδά δηλαδή. Το πρώτο είναι τι αντίδραση υπάρχει αυτή τη στιγμή και τι είδους κρίση τι είδου κρίση υπάρχει σε σχέση με το Ιράν και την κατάρριψη του αεροσκάφους που, ε, στην οποία προέβη πριν από κάποιες εβδομάδες. Δεύτερον, και εσείς μιλήσατε και είναι πολύ σημαντικές οι σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυβέρνησης Καναδά όσον αφορά την ηθαγένεια. Όχι δηλαδή μόνο το τι, ποιος κυβερνά, αλλά και το, τους πολίτες. Σε σχέση με τις τελευταίες συνθήκες που έχουν υπογραφεί ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Καναδά θα υπάρχει, ε, είστε θετικοί ή περισσότερο ε, υποδεικνύονται οι αντιπαραθέσεις ε, μεταξύ των δύο πλευρών της στρατηγικής, όσον αφορά δηλαδή τη στρατηγική εμπορική συμφωνία και τη ΣΥΤΑ. Ευχαριστώ πολύ. Γιόλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και την ε, πρέσβυρα για μια πολύ περιεκτική παρουσίαση της κατάστασης. Ήδη μιλήσατε για τις αυξημένες εμπορικές συναλλαγές, αλλά αυτό είναι ένα καλό ε, μήνυμα και προς τα κράτη-μέλη μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά. Μιλήσατε και για τη Γεωργία. Πλην αυτής, ποιοι άλλοι τομείς παρουσιάζουν αύξηση των εμπορικών συναλλαγών. Αν δεν μπορείτε να μου δώσετε τώρα τα νούμερα, γραπτός ε, θα ήθελα να λάβω μια απάντηση. Στην Αρκτική επίσης, τι γίνεται. Διότι υπάρχει επιθετικότητα της τάσης της Ρωσίας. Ε, δεν ξέρω αν ε, έχετε κάποια νέα για το κατά πόσον θεωρείτε ζήτημα αυτό ακόμη για τον Καναδά. Τι πιστεύει η κοινή γνώμη και ποιες είναι επίσης ε, και οι συνοκαναδικές σχέσεις ε, όταν πριν από 13 μήνες ε, υπήρξε η σύλληψη της Κερασουέ και η Huawei βέβαια είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. δεν ξέρω αν μπορείτε να μας πείτε τίποτε τι θα γίνει με αυτή την εταιρεία και σε σχέση και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι θα γίνει με τα αιτήματα ή τις απαιτήσει των Κινέζων ξέροντας ότι στο Δυτικό Ειρηνικό υπάρχουν, υπάρχει ένα μεγάλος πληθυσμός και πώς θα το αντιμετωπίσετε και αυτό τέλος. Ξέρω ότι στην Ανατολική Ευρώπη, ιδίω στην Ουκρανία, υπάρχει έντονη παρέμβαση, μάλλον ε, δραστηριοποίηση του Καναδά, γιατί υπάρχει και καναδική διασπορά εκεί και θα ήθελα να μας πείτε λίγο περισσότερες ε, λεπτομέρειες για τις συγκεκριμένες δράσεις, αν ε, γνωρίζετε κάτι, θα αναλυφθεί από τους ε, Καναδούς, είτε στην Ουκρανία, είτε σε κάποια άλλη χώρα της Ανατολικής Γειτονίας. Ευχαριστώ. Μωρένο Σάνσεφ. Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και την ε, κυρία Χέρντα. Εγώ είμαι και εισηγητής μόνιμος εισηγητής για την Συμφωνία ΣΥΤΑ εκ του Κοινοβουλίου. Είμαι και αντιπρόεδρος τη Αντιπροσωπείας για τη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Καναδά, άρα δεν παρεμβαίνω μόνο ω μέλο αυτή τη επιτροπή. Είπατε κι εσεί ότι ο Καναδά ίσω είναι η πιο ευρωπαϊκή χώρα εκτό Ένωση. Και συμφωνούμε. Ε, έχουμε πολλέ κοινέ αξίε ε, και πολλά κοινά προβλήματα. Αυτή η συμφωνία, η ΣΕΤΑ, το είπε και η κυρία είναι πολύ περισσότερο από εμπορική συμφωνία. Μιλήσατε για τη μετανάστευση, για την κλιματική αλλαγή, την ισότητα μεταξύ των φύλων και νομίζω ότι εκεί πρέπει να ε, εργαστούμε. Είπατε ότι δεν υπάρχει μεγάλη αλλαγή ε, στον Καναδά, λίγο πολύ η σύνθεση της κυβέρνησης είναι ίδια και νομίζω ότι και εμείς θα κάνουμε ότι μπορούμε για να μην υπάρξουν αλλαγές ούτε από την πλευρά μας. Μια ερώτηση, πώς βλέπετε τη διαδικασία κύρωσης. Ορισμένες χώρες ε, έχουν κάποιες επιφυλάξεις όπως γνωρίζουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Διότι πολλές φορές υπάρχει παραπληροφόρηση. Εμείς τι πληροφόρηση μπορούμε να δώσουμε γιατί σε τελική ανάλυση τα κοινοβούλια είναι κυρίαρχα και αυτά θα ψηφίσουν. ότι όμως δεν έχουν όλες τις πληροφορίες. Μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε κάτι να κάνουμε από πλευράς κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Να προσθέσω κι εγώ, αν μου επιτρέπετε, ένα ερώτημα. Το 40% περίπου των εμπορικών συναλλαγών της Ένωσης με τον Καναδά ήταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, που τώρα είναι εκτός ήταν ένα είδος πύλης ε, κοινοπολιτεία και τις είπα και άλλες χώρες ε, το Ηνωμένο Βασίλειο τώρα που είναι εκτό Ένωσης τι περιμένουμε βλέπουμε κάτι ήδη βλέπουμε μια μετατόπιση ενδεχομένω εταιριών ε, οι έδρε μεταφέρονται σε άλλες ε, χώρες τι γίνεται Υπάρχει ακόμη μια στάση αναμονής μέχρι ότου έχουν ή εταίροι κάποια ιδέα για τη μελλοντική μας συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Αν δεν θέλουν άλλοι έρθουν το λόγο, έχετε εσείς κυρία Πρέσβη το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσω από το τέλος. ΣΕΤΑ, επικύρωση, εμπόριο και πώς ε, διαγράφεται η κατάσταση από εδώ και πέρα. Να σας επαναλάβω ότι βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο με την ε, Αγγλία, με την ε, Βρετανία για ένα ακόμη χρόνο. Δεν θα αλλάξουν πολλά. Η Βρετανία βέβαια θα πρέπει να διαπραγματευτεί αν έχει ενδιαφέρον και συμφέρον και ξέρουμε ότι έχει, να έχει ίσως και μια εμπορική συμφωνία με τον Καναδά. Εμείς προς το παρόν εκτιμούμε και εξολογούμε την κατάσταση, μελετούμε τα στατιστικά στοιχεία, για να δούμε αυτό τι σημαίνει για εμάς. Και δεν ε, αφορά αυτό μόνο τον Καναδά, είναι μια γενική τάση. Για το εμπόριο, τις εξελίξεις, ε, τι θα γίνει χωρίς την παρουσία των ε, Βρετανών, τα ξέρετε πολύ καλά. Και σίγουρα συζητείτε επί αυτό το θέμα και το έχετε ήδη συζητήσει. Εμείς στην ΕΕΔ που είμαστε και αρμόδιοι για τη σχέση με τις τρίτες χώρες, ακριβώς το ίδιο κάνουμε. Δηλαδή μελετούμε την κατάσταση προς το παρόν για να δούμε αν χρειάζεται ένας επαναπροσανατολισμός και βέβαια βλέπουμε ότι ήταν ε, πολύ στενές επαφές των Βρετανών με την καναδική κυβέρνηση. Αυτό το βλέπει κανείς και στους δικούς μου τομείς αρμοδιότητα, Ήδη έχουν υπογράψει μάλιστα κάποιες συμφωνίες με τρίτες χώρες. Άρα εξαρτάται από αυτούς. Δεν έχω νούμερα να σας δώσω. Οι συνάδελφοι μου από την Εμπόριο και όχι εμείς από την ΕΕΔ μπορούμε να σας δώσουμε αυτά τα στοιχεία. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε για τη ΣΕΤΑ και θα το κάνουμε και ήδη έχουμε ξεκινήσει είναι να δίνουμε χέρα βοηθείας προς τους συναδέλφους από την Γαμαδελτά Εμπόριο για να δουν, να τους εξηγήσουμε γιατί η ΣΕΤΑ και η SPA είναι σημαντικές συμφωνίες. Μιλούμε με τα κράτη-μέλη, βοηθούμε και με την ενημερωτική εκστρατεία. Να δούμε ποια ήταν τα ωφέλη αυτών των δύο συμφωνιών. Πραγματικά τον 1,5 χρόνο που ισχύει αυτή η συμφωνία. Ήταν πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον της άλλης πλευράς. Ε, υπήρχαν ε, διάφορες εκδηλώσεις, συμμετείχαν και αυξάνεται το ενδιαφέρον. Είχαμε και κάποιες διμερείς ομάδες εργασίας. 27 είναι τώρα στον αριθμό και αυξάνονται. Οι εμπειρογνώμονές μας θέλουν να έρθουν σε επαφή με τους ομολόγους τους και βλέπουμε πραγματικά να υπάρχει περιθώριο ανάπτυξης μιας ε, πολύ καλής ε, ευρεία σχέσεως. Και όχι μόνο ο αριθμός των ομάδων εργασίας είναι μεγάλος, αλλά υπάρχουν και σημαντικές ε, και πολλές συναντήσεις, ανταλλαγές απόψεων. Δεν είναι κάτι θεωρητικό που μένει στα χαρτιά. Αντίθετα, έρχονται όλο και περισσότερο σε μας Για την ε, ΣΕΤΑ, όπως σας είπα, θα εργαστούμε μαζί με τα κράτη-μέλη για να δούμε τι μπορεί να βοηθήσει και γνωρίζουμε πως ο Καναδάς και οι καναδικές πρεσβείες ε, δραστηριοποιούνται τα μάλα και στα κράτη-μέλη για τον ίδιο σκοπό. Έρχομαι στην Ουκρανία. Η διασπορά είναι πολυάριθμη, είναι πολυπληθής προηγούμενη κυβέρνηση Τριντό ε, βοήθησε πολύ και με τις μεταρρυθμίσεις στην Ουκρανία είχαν έντονη δράση, προσπάθησαν να βοηθήσουν και με την έκρηση αφόρων νομοσχεδίων για τον παρόνομο πλουτισμό, διαφθορά κτλ. Και έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Έχουμε καλό συντονισμό με τον Καναδά. ιδίω στην Ουκρανία και σε πολλά ζητήματα. Θέλουμε να υπάρχει συνέργεια και να έχουμε μία παράλληλη συντονισμένη δράση. Προς τώρα, στην Αρκτική, Ξέρετε ότι υπάρχει δικό σα απεσταμένο τη ΕΕ για την Αρκτική. Ανοίγει ένα νέο χώρο, λοιπόν, μια νέα περιοχή για εμά. Η ομάδα για την Αρκτική δυστυχώ δεν περιλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Αρκτικό Συμβούλιο. Κάποια κράτη-μέλη ναι, αλλά η πολιτική μα ουσιαστικά είναι αρκετά συντονισμένη με αυτήν τον Καναδά και έχουμε και τακτικέ συναντήσει με τον Καναδά για την Αρκτική συγκρίνουμε τις πολιτικές ε, και καθορίζουμε τις προτεραιότητές μας. Παρακολουθούμε ε, τη δράση των ε, κρατών μελών και βλέπουμε ποιες είναι και οι προτεραιότητες των Καναδών και πώς αυτές συνδυάζονται με αυτές των κρατών μελών. Βέβαια, είναι λογικό να είναι διαφορετικές προτεραιότητες. Αυτό πάντοτε συμβαίνει. Τώρα, τι κάνει η Ρωσία στην Αρκτική, το γνωρίζουμε, παρακολουθούμε βεβαίως την κατάσταση και μάλιστα από πολύ κοντά. Όλοι πρέπει να συνεργαστούμε σε αυτή την περιοχή. Να παραμείνω στα της εξωτερικής πολιτικής ε, και να περάσω στην Κίνα. Κίνα όπως και η Ουκρανία αυτές είναι οι δύο προτεραιότητες ε, για τις οποίες είχαμε πολύ συντονισμό, πολύ μεγάλο συντονισμό με την καναδική πλευρά τα τελευταία χρόνια. Η Καναδί ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένη με την ε, δράση μας, με την υποστήριξη που τους παρήχαμε. Ιδίω σε σχέση με το άτομο το οποίο κρατεί στην Κίνα, στην Κίνα. Και οι διπλωματικές μας ε, προσπάθειες, ελπίζω, θα βοηθήσουν την απελευθέρωση τα ατόμα αυτό στο μόνο δυνατό. Είναι βέβαια λεπτό θέμα, διμερές, ε, παρόλα αυτά αν μπορούμε να βοηθήσουμε πάντοτε το προσπαθούμε. Γιατί τελικά πρόκειται για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει να είναι σεβαστά. Υποστήριξη για τη ΣΥΤΑ. Ναι, υπήρξε αρχικά κάποια αντίσταση και κάποιες κριτικές, αλλά νομίζω ότι με τα νέα στοιχεία τα οποία βλέπω το φως της δημοσιότητας, η αντίθεση και αντίδραση, όχι στον Καναδά, αλλά και εδώ στην Ευρώπη σε βάρος της ε, ΣΕΤΑ, μειώνεται γιατί υπάρχει κατανόηση πλέον της σημασίας αυτής της συμφωνίας ότι τα ωφέλη και για την Ευρώπη και για τον Καναδά είναι μεγάλα και πολλά. Άρα δεν βλέπουμε πλέον τόσο έντονες επικρίσεις τον τελευταίο καιρό. Ακριβώς λόγω του ότι προσπαθούμε να προβάλλουμε καλά επιχείρηματα και καλά παραδείγματα σε αυτή τη συζήτηση. Υπήρξε και ένα ερώτημα για την πρόσφατη κατάσταση. Υπάρχουν ψηφίσματα. Υπάρχει ψήφισμα ε, του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο Καναδάς που θέλει να είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας στηρίζει. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε το Ιράν. Υπάρχουν κάποια περιθώρια. Γενικώ ομονοούμε νομίζω με τους εταίρους μας πάνω σε αυτά τα θέματα. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν συνάδελφοι που θα ήθελα να θέσουν ίσως κάποιο ερώτημα. Αν όχι, να σας ευχαριστήσω που ήρθατε εδώ. Συνεχίστε να παρακολουθείτε την κατάσταση για να μπορείτε να μας ενημερώνετε όποτε το επιθυμούμε. Σας ευχαριστώ. Βεβαίως θα είναι χαρά μου. Colleagues, we have an eight-minute break. Από τη θα κάνουμε 8 λεπτά διάλειμμα. Γιατί ο Επίτροπος θα έρθει 4 και 4. Και θα είναι και κλεισμένο των ε, θηρών οι συνεδρίες από εδώ και πέρα. Όλοι αυτοί οι νέοι λοιπόν που όμως δεν έχουν κάποια επίσημη ιδιότητα στην ομάδα ή δεν είναι βουλευτές, όλοι αυτοί οι πολύ ωραίοι νεαροί και νεαρές δυστυχώς να αποβιβαστούν.